Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση. Να ενημερώσω τον Νίκο ότι σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 δεν ζητήθηκε να ψηφίσουμε τα διορθωτικά που ανακοινώθηκαν χθες στις 5 το απόγευμα, οπότε τα διορθωτικά θεωρούνται ως εγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.